Μετά λοιπόν από 27 χρόνια της ισόβιας κάθριξης ε, που του είχε ε, αγορευτεί το 1984. Ο κύριος Μαντέλα έχει επίσης ε, κερδίσει το βραφείο Ζαχάροφ το 1988 όταν θεσμοθετήθηκε το βραβείο αυτό. Ο Γέρζι Μπούζεκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ευκαιρία αυτή είπε «Ο Νέλσον Μαντέλα αποτελεί έμπνευση ε, για όλους ε, και μένει χαραγμένος βαθιά στην καρδιά και στην ψυχή όλων των ανθρώπων της Αφρικής αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Το όνομα του Νέλσον Μαντέλα θα είναι άρρηκτα ε, συνδεδεμένα στο με τον αγώνα για την ελευθερία και την δημοκρατία. Ο Νέλσον Μαντέλα πρόκειται, ε, ε, απεικονίζει την ακεραιότητα στην πολιτική ε, ζωή και επίσης σηματοδοτεί την αρχή της συμφιλίωσης ανάμεσα σε παλιούς εχθρούς και αποτελεί έμπνευση για το μέλλον. Ο συνεχής αγώνας του Νέλσον Μαντέλα και η προσπάθειά του να καταπολεμηθεί ο ιός του AIDS σημαίνει ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κούσμαν. Κύριε Κούσμαν, παρακαλώ, ως πρόεδρο τη Αντιπροσωπείας με την Νότια Αφρική. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, γιατί ξέρω ότι όλοι έχουμε άλλε ασχολίες να κάνουμε. Πριν από 20 χρόνια ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίστηκε μετά από 27 χρόνια πολιτικού ε, εγκλισμού. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι για το δρόμο του προς την ελευθερία. Ήταν μια μέρα που άλλαξε την ε, Νότια Αφρική. Τότε ε, τέθηκαν τα θεμέλια για μια σύγχρονη Νότια Αφρική που θα ξεχνούσε την οργή και το μίσος. Ο Νέλσον Μαντέλα είναι, κύριε Πρόεδρε, ε, κατά την άποψή μου, ένα ζωντανό σύμβολο και με την απελευθέρωσή του απελευθέρωσε την χώρα του και έριξε στο σκουπεδοτενικέ της ιστορίας ε, το apartheid και δημιούργησε μια πολυφιλετική δημοκρατία στη Νότια Αφρική. Τον χαιρετίζουμε λοιπόν.